να ανακάμψουμε, να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία και ανταγωνιστικότητα και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Κύριε Επίτροπε Βαρνιέ, με την παρουσίαση αυτή ολοκληρώθηκε η συζήτηση και περνάμε ευθύ αμέσως στο επόμενο θέμα που είναι οι συμπράξεις καινοτομίας. Είναι προφορική ερώτηση. Πρώτα απ' όλα θα δώσουμε το λόγο στους συντάκτες της προφορικής αυτής ερώτησης με πρώτη την κυρία Μέρκης που έχει δύο λεπτά στη διάθεσή της. Παρακαλώ, κυρία Μέρκης. Κύριε Πρόεδρε, το 90% του κόσμου πιστεύει ότι η καινοταμία μπορεί να βοηθήσει να έχουμε μια καλύτερη οικονομία. Συμφωνούμε. Όμως, επίγει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει αποφασίσει να συζητήσουμε τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο που μας έρχεται για αυτά τα θέματα. Γιατί δεν είναι μια μεγάλη πρόκληση. Έχουν λυθεί όλες οι προκλήσεις. Το θέμα της γύρασης του πληθυσμού για παράδειγμα. Όχι. Γι' αυτό λοιπόν είναι αναγκαίο να συζητήσουμε τα θέματα της καινοτομίας όσο γίνεται πιο γρήγορα. Τι είναι οι συμπράξεις καινοτομίας. Παραμένει ανοιχτό κάπως το ζήτημα. Δεν θέλουμε ένα νέο όργανο, το είχαμε πει αυτό, αλλά θέλουμε κάτι καλύτερο. Και σημαντικό είναι μακροπρόθεσμα να δώσει αποτελέσματα, να είναι ένα μέσο το οποίο θα λειτουργήσει καλά εν ώψη του 2020. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι οι συμπράξεις καινοτομία πρέπει να είναι κάτι συγκεκριμένο τεχνολογικά ουδέτερο και κοντά στην αγορά και με συγκεκριμένες προθεσμίες και με τη συμμετοχή όλων των σημαντικών εταίρων και της βιομηχανίας και της κυβέρνησης και της κοινωνίας των πολιτών που αποτελούν και τη βάση στο κάτω-κάτω της καινοτομίας. Είναι πολύ καλό που βασιζόμαστε στην, ε, στους πολίτες οι οποίοι θα φροντίσουν να αντιμετωπιστεί και το θέμα της γύρανσης του πληθυσμού. Όλες οι συμπράξεις καινοτομία πρέπει να είναι αποτελεσματικές, να αποτελούν μια πηγή και μετά βέβαια υπάρχει και το θέμα της ε, ενέργειας και εκεί που χρειάζεται καινοτομία. Το Συμβούλιο πρέπει να βοηθήσει με ενθουσιασμό. Είναι αναγκαίο. Δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Η οικονομία δεν είναι μόνο το ευρώ, δεν είναι μόνο το σύμφωνο σταθερότητα, είναι η απασχόληση, είναι η καλύτερη θέση τη Ευρώπη μέσα στον κόσμο και αν δεν έχουμε καινοτομία, πώ θα το πετύχουμε αυτό αλλιώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η Αμάλια Σαρτόρη έχει τώρα το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Η πρόταση της Κομισιόν που περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση Ένωση της Καινοτομίας που υιοθετήθηκε στις 6 Οκτωβρίου είναι αναπόσπαστο τμήμα της ε, στρατηγικής για το 2020. Η πρωτοβουλία αυτή θέλει να αποτελέσει μια συγκεκριμένη αποτελεσματική και βιώσιμη απάντηση στα κύρια προβλήματα της κοινωνίας μας. Ανάμεσα στις διάφορες ε, προτάσεις ε, που γίνονται μέσα σε αυτή την απόπειρα να δοθεί ζωή σε μια πραγματική ένωση της καινοτομίας, ένα από τα πιο καινοτόμα στοιχεία αντιπροσωπεύεται από αυτές τις ε, συμπράξεις καινοτομίας με στόχο την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων είναι απαραίτητο να επιλεγούν ίσως τέσσερα αυτές ε, συμπράξεις ε, και για αυτό το στόχο έχει εντοπίσει η Κομισιόν ορισμένες συγκεκριμένες προκλήσεις που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει η κοινωνία μας στις επόμενες δεκαετίες. Σε σχέση με αυτές τις καινοτόμια, το Ευρωκοινοβούλιο επέλεξε να εκφράσει αντίθεση Εγώ είμαι η για το ΕΛΚ για το συγκεκριμένο ψήφισμα και μετά από σύντομε διαπραγματεύσει όλε οι πολιτικέ ομάδε υπέγραψαν ένα ψήφισμα για το οποίο δεν υπάρχουν προβλήματα. Θέλω να, υπογραμμίσω ότι η δική μα συμβολή ήταν ε, ουσιώδη έτσι ώστε να επιτύχουμε ότι οι δύο συμπράξει που θα ξεκινήσουν μετά από την πιλωτική πρωτοβουλία για την ε, γύρανση με καλή υγεία θα απαιτήσουν ευφυείς λύσεις ώστε να στηρίξουν σε διάφορες πόλεις ε, της Ευρώπης ε, προηγμένα προγράμματα που στόχο έχουν να στηρίξουν ε, τους στόχους του 2020 και τις πρώτες ύλες τις μη ενεργειακές ώστε να δοθούν απαντήσεις στα μεγάλα και δύσκολα προβλήματα που ενδιαφέρουν την κοινωνία μας σε αυτό το πλαίσιο. Τους επόμενους μήνες μια ομάδα εργασίας εσωτερικής στην Κομισιόν θα αποφασίσει στις λεπτομέρειες της, της κυβέρνησης, της χρηματοδότησης, του προπολογισμού αυτών των πρωτοβουλειών που θα ξεκινήσουν με την πρώτη σύμπραξη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ το... Ο Γιώργος Χατζημαρκάκης. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τι κάνει η πολιτική καινοτομία της Ευρώπης και η πολιτική έρευνα της Ευρώπης. Αν θέσουμε αυτό το ερώτημα ε, στον μέσο Ευρωπαίο στο δρόμο δεν θα μας δώσει μία σαφή ε, απάντηση διότι δεν ξέρει την προστιθέμενη αξία της καινοτομία και της έρευνας στην Ευρώπη. Γι' αυτό χαιρετίζουμε ε, την πρόταση αυτή η οποία καθορίζει τι σημαίνει καινοτομία. Δηλαδή να κάνουμε κάτι από νέο ένα προϊόν, ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, από ε, τίποτα. Και θα πρέπει να το καταλάβει και ο πολίτης για να καταλάβει τι κάνουμε με τα χρήματα του ο Ευρωπαίος Ορολογούμενος Έχουμε λοιπόν ακόμη δύο χρόνια τα οποία προσπαθούμε να προσθέσουμε στην υγιή διαβίωση και γι' αυτό ε, σας ευχαριστώ διότι αυτή η συνεργασία αποβλέπει σε αυτή την ε, δράση, δηλαδή να υπάρξει καινοτομία και γι' αυτό σας στηρίζουμε. Θέλω όμως να πω ότι ε, οι συγητές και οι προλαλοί σας ανέφεραν, εάν δούμε τα τωρινά, ε, τις τωρινές δυνατότητες, τα kicks, τα jetties, τα innovation, Innovation Programs, δηλαδή προγράμματα τα οποία ήδη υπάρχουν όπως και το SIP. Εάν προσθέσουμε και άλλο νέο πρόγραμμα θα είναι αδιαφανές το σύνολο και γι' αυτό οι συνεργασίες και ενοτομίες θα πρέπει να συμβάλλουν να υπάρξει ένα συνολικό σύνολο και αυτό θα είναι μόνο αποδεκτό εάν είναι σαφές για το φορολογούμενο. Να είναι σαφές ότι προσθέτει η ευχαριστημένοι. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τοσινόφσκι για δύο λεπτά. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η πρωτοβουλία της Επιτροπής να δημιουργήσει πειραματικά προγράμματα όσον αφορά τις συμπράξεις καινοτομίας με τίτλο «Ενεργά και γη γυρατιά» είναι κάτι πολύ αξιόλογο. Η επιλογή δείχνει πως ε, είναι δύσκολο να καταλήξουμε σε αποφάσεις και να χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένα κριτήρια. Οι διάφορες πρωτοβουλίες είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Έπειτα υπάρχουν διαφορετικές νοτροπίες, διαφορετικές ιστορικές παραδόσεις, διαφορετικές προσεγγίσεις από τα κράτη-μέλη. Οπότε είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πόσο καινοτόμα θα είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να λύσει αυτό το πρόβλημα της επιλογής. Ελπίζω τα κριτήρια δεν θα βασίζονται σε μια γενική μόνο περιγραφή, αλλά ότι η Επιτροπή θα δώσει πραγματική βοήθεια. Από την εμπειρία που έχουμε εμείς μέχρι τώρα, βλέπουμε ότι υπάρχουν και προτάσεις και για τις έξυπνες πόλεις και για τις πρώτες ύλες. Αν σκεφτούμε τι, τι προβλήματα θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον, νομίζω ότι πρέπει να προτιμήσουμε τις πρώτες ύλε. Σήμερα και στο εγγύς μέλλον πάρα πολλές χώρες θα βρεθούν υπό μεγάλη πίεση για να έχουν υλικά για την ενέργεια και τη βιομηχανία. Πολλοί το έχουν καταλάβει αυτό ήδη. Πρέπει να βρούμε νέα, νέες πηγές κάτι πολύ βασικό για τη μελλοντική μας ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά και αυτό θα επηρεάσει και πολλούς άλλους τομείς και τις κοινωνικές πτυχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και οι κανόνες πρέπει να είναι ξεκάθαροι και να φροντίσουμε ότι θα υπάρχει πρόσβαση στα νέα υλικά, γιατί είναι αυτό το στοίχημα του μέλλοντος. Ευχαριστούμε. Να τηρείτε το χρόνο σας παρακαλώ. Μαρίσα Ματίας τώρα παρακαλώ που είναι συντάκτρια και αυτή της ερώτησης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Περί ενός από τα θέματα που είναι μία από τις κύριες προτεραιότητές μας συζητάμε σήμερα για την πολιτική καινοτομία. Και νομίζουμε ότι μπορεί με τις εταιρικέ σχέσεις για την καινοτομία να προωθηθεί το θέμα αυτό και το σχέδιο έκθεση που συζητούμε εδώ έχει να κάνει με τα θέματα αυτά. Είναι πολλά ακόμα τα οποία πρέπει να αναφερθούν επίσης σε ό,τι αφορά τα μελλοντικά σχέδια και σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες. Ποιος θα καθορίσει τις προτεραιότητες και με ποια κριτήρια. Και εδώ υπάρχουν ακόμα αμφιβολίες. Εγώ όμω θέλω να κάνω ορισμένες παρατηρήσει συγκεκριμένε σε σχέση με αυτό το πρώτο σχέδιο για την ενεργή γύρανση και νομίζω ότι προφανώς αυτά τα πράγματα πρέπει να έχουν ένα θετικό χαρακτήρα και να εστιάσουμε καλύτερα σε ένα τμήμα του πληθυσμού το οποίο είναι όλο και πιο ευάλωτο και βρίσκεται όλο και σε πιο μειονεκτική θέση στην Ευρώπη. Είναι απαραίτητο όμως να προσθέσουμε και μερικά ακόμα ερωτήματα. Μου φαίνεται ότι είναι κάπως αντιφατικό να παρουσιάζεται ένα σχέδιο στον τομέα αυτό τη στιγμή που εμείς ζητάμε να ενισχύσουμε την καινοτομία. Αν θέλουμε να έχουμε μια καινοτομία βιώσιμη στο πλαίσιο αυτό, δεν μπορούμε να την έχουμε να συνάδει με μια συνεχή επίθεση εναντίον αυτού του στρώματος του πληθυσμού που υφίσταται συνεχείς περικοπές που ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης επίσης υφίσταται μεγάλες πιέσεις, μειώνονται οι δημόσιες δαπάνες και οι επενδύσεις. Δεν μπορούμε αυτά να τα συμβιβάσουμε με μια πολιτική που θέλει να έχει μια φιλόδοξη αντιμετώπιση για την ενεργό ε, γύρανση. Θεωρούμε λοιπόν ότι εδώ υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση με τα μέτρα ε, λιτότητος και τις περικοπές που γίνονται στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Μέσης. Θέλουμε να έχουμε πολιτικές οι οποίες δεν θα είναι απλώς πολιτικές λιτότητος, αλλά που θα είναι πολιτικές οι οποίες θα βοηθούν την αγορά εργασίας και θα δίνουν δυνατότητες και διεξόδους στον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο Πρόεδρος. Και τώρα, ο κύριος ο Υπουργός ξέρεξε. έχει το λόγο. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, εκ μέρους του Συμβουλίου. Έχετε το λόγο. Euh, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, Χαίρομαι πολύ που μας δίνεται η ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί για την πρωτοβουλία αυτή φάρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καινοτομία και ιδιαίτερα για την νέα αυτή ιδέα της σύμπραξης καινοτομίας. Είναι σίγουρα ένα στοιχείο κλειδί της ανακοίνωσης που παρουσίασε αρχές Οκτωβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εννοείται ότι στο στάδιο αυτό το Συμβούλιο εξετάζει το θέμα. Ετοιμάζουμε τα συμπεράσματά μας για το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της 26 Νοεμβρίου. Όπως θα θυμόσαστε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 17 Ιουνίου ολοκλήρωσε την εκπόνηση της στρατηγικής 2020. Εκεί καθορίζονται μεγάλοι στόχοι που είναι να βελτιωθούν οι συνθήκες έρευνας και ανάπτυξης προκειμένου όλος ιδιαιτέρως να δώσουμε 3% του ΑΕΠ σαν επενδύσεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα προς αυτούς τους τομείς. Προσωπικά πιστεύω ότι θα είναι δύσκολο να φανταστούμε λιγότερο από 3% που ήδη αναφέρονται στη στρατηγική της Λισαβόνας και ότι τώρα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να τα καταφέρουμε. Η πρωτοβουλία αυτή λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καινοτομία που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθορίζεται από αυτόν ακριβώς το στόχο. Και το Συμβούλιο θέλει με ιδιαίτερη προσοχή να εξετάσει το θέμα το Συμβούλιο είχε μια πρώτη άτυπη ανταλλαγή απόψεων τον Ιούλιο που μας πέρασε επ' αυτού και στη συνέχεια επίσημα στις 12 Οκτωβρίου που μας πέρασε. Μετά από αυτή τη συζήτηση η Προεδρία κατέληξε σε ένα σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου που εξετάζεται αυτή την εποχή και είναι στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 25ης και 26ης Νοεμβρίου που μας έρχεται. Υπογραμμίζω εδώ ότι η Προεδρία φρόντισε η έρευνα και η βιομηχανία, οι δύο αυτοί τομείς, να συνεργάζονται σε αυτό το φάκελο. Με εξαίρετα αποτελέσματα. Εξάλλου το Συμβούλιο που μας πέρασε είχαμε από κοινού Συμβούλιο και πρέπει τώρα να καταλήξουν από κοινού σε συμπεράσματα τέλη Νοεμβρίου. Εξάλλου, η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως και οι εργασίες του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας, θα τροφοδοτήσουν την προετοιμασία της συζήτησης που θα γίνει για την έρευνα και την καινοτομία που θα γίνει μέχρι τα τέλη της χρονιάς στο Συμβούλιο. Ανταλαμβάνεστε δηλαδή πόσο μεγάλη σημασία έχουν αυτά τα θέματα για τους επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων στο Συμβούλιο. Εγώ πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικό στο τι λέω μέχρι να αποφανθούν αυτοί. Πάντως, επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω ότι το θέμα της καινοτομία ή πιο σωστά το τρίγωνο της γνώσης με την ευρύτερη έννοια εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία δηλαδή. Το τρίγωνο λοιπόν αυτό δεν είναι κάτι νέο ούτε για το Συμβούλιο ούτε για το Κοινοβούλιο. Από πλευράς του Συμβουλίου, σε ένα γενικότερο πλαίσιο για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνα, το θέμα αυτό τακτικά βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητα. Για παράδειγμα, ε, το όραμα 2020 για το χώρο έρευνας του Σεπτεμβρίου του 2008 και πιο πρόσφατα στα συμπεράσματα του Συμβουλίου που λέει να δημιουργήσουμε μια καινοτόμα Ευρώπη που εγκρίθηκε το Μάιο που μας πέρασε υπό Ισπανική Προεδρία. Και μπορώ εδώ να αναφέρω χωρίς να καλύπτω όλο το θέμα τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Πρώτα απ' όλα, οι πρωτοβουλίες θα πρέπει να έχουν να κάνουν με κάθε μορφή καινοτομία στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Δεύτερο στοιχείο. Πρέπει να θέσουμε τις βάσεις για μια πιο αποτελεσματική χρηματοδότηση όσον αφορά την ανάπτυξη και την καινοτομία. Τρίτον, οι δημόσιες αγορές ναι. που δεν έχουν εκμεταλλευτεί πλήρως ακόμα πρέπει να στηρίξουν την καινοτομία ναι. για ένα προϊόν λοιπόν και για τις υπηρεσίες. Τέταρτον, οι μη τεχνολογικές καινοτομίες και στον τομέα του design, των υπηρεσιών και της πολιτιστικής δημιουργίας αποτελούν επίσης σημαντικούς τομείς. Πέμπτον, η εκμετάλλευση των προσπαθειών που γίνονται στην έρευνα είναι κάτι που απαιτεί διαχείριση και προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, αποτελεσματική μάλιστα, όπως επίσης και διάδοση της καινοτομίας. Τέλος, οι πολιτικές και τα προγράμματα σε θέματα ανάπτυξης και έρευνας και τα μέσα που τα συνοδεύουν πρέπει να απλοποιηθούν και να εξαρθολογιστούν. Και χαίρομαι εδώ που υπάρχει σύγκληση απόψεων με την, Ευρωπα... με την Επιτροπή, την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ήτρε, και το βλέπουμε αυτό στην έκθεση της κυρίας Καρβάλιο. Οι συμπράξεις καινοτομία δεν πρέπει να περιπλέξουν ακόμα περισσότερο τα πράγματα, αλλά αντίθετα πρέπει να συμμετέχουν στην απλοποίηση. Η περιφερειακή διάσταση είναι εξάλλου πάρα πολύ σημαντική για την καινοτομία και σχετικά η ευρωπαϊκή πολιτική καινοτομίας θα πρέπει να υποστηρίξει όλου αυτού οι οποίοι είναι σημαντικοί φορεί καινοτομία, ιδίω οι μικρομεσαίες επιχειρήσει που θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερη υποστηρίξη σε περιφερειακό επίπεδο. Ο ανθρώπινο παράγων είναι στην καρδιά τη έρευνα και τη καινοτομία. Η Ευρώπη θα πρέπει να ενισχύσει την ικανότητά τη, να διατηρήσει το επιστημονικό της κεφάλαιο και να προσελκύσει ταλέντο από τρίτες χώρες. Μετά από αυτές τις σκέψεις που είναι γενικού χαρακτήρα, θα ήθελα να απαντήσω στα τέσσερα πιο συγκεκριμένα και απτά ερωτήματα τα οποία έχετε θέσει. Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ζητημάτων, των θεμάτων μάλλον, για την εταιρική σχέση και την καινοτομία, ακόμα και αν το Συμβούλιο δεν έχει μου φαίνεται ότι είναι ομόφωνο στο ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με πιλωτικού χαρακτήρα πρωτοβουλίες. Και η Κομισιόν πρότεινε να ξεκινήσει αυτή την πιλωτική πρωτοβουλία για την γύρανση ξεκινώντας από το 2011 και περιλαμβάνει και μια σειρά άλλων θεμάτων για τα οποία είναι έτοιμη η Κομισιόν να καταθέσει προτάσεις το 2011 και κάποια από εσά έχετε υποστηρίξει αυτές τις ιδέες. Εξορισμού εξάλλου ένα πιλωτικό σχέδιο έχει πειραματικό χαρακτήρα και χωρίς φυσικά να περιμένει όλες οι προϋποθέσεις να πληρούνται. η επιλογή των θεμάτων για τις μελλοντικέ εταιρικές σχέσεις είναι ένα από τα μείζωνα θέματα τα οποία είναι υποσυζήτηση στους κόλπους του Συμβουλίου. Και σας υπενθυμίζω την άσκηση κοινού προγραμματισμού της έρευνας στην Ευρώπη για να απαντήσουμε στις κύριες προκλήσεις της κοινωνίας <clears throat> που ξεκίνησε από το Συμβούλιο το 2008. Και με την ευκαιρία αυτή τα κριτήρια τα οποία θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα και στο πλαίσιο της εταιρική σχέσης για την καινοτομία είχαν ήδη θεσπιστεί. Η ευρύτητα της πρόκλησης αυτής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ανάγκη μιας πλήρους δέσμευσης και προσήλωσης των εμπλεκομένων, η προστιθέμενη αξία, η ανάγκη να μεταφράσουμε την καινοτομία σε ωφέλη για τον Ευρωπαίο πολίτη και για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Ατενίζω λοιπόν μια ευρεία σύγκληση μεταξύ των προηγουμένων προσεγγίσεων του Συμβουλίου και των γενικών προϋποθέσεων που προτείνει η Κομισιόν μέσα στην ανακοίνωσή της. Και εξ άλλου, <clears throat> στις συζητήσεις που είχαμε μέχρι τώρα, οι συνάδελφοί μου τόνισαν ιδιαίτερα την ανάγκη να έχουμε μια προσέγγιση η οποία είναι μια ανερχόμενη ε, προσέγγιση να υπάρξει απλότητα, ελαφρότητα των δομών, συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, ιδίως τις μικρές αλλά και τις μεσαίες επιχειρήσεις και επίσης την βελτιστοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων που υπάρχουν ήδη. Έρχομαι τώρα στο χρονοδιάγραμμα και στην αρχή της ευκυβερνησίας, που είναι <clears throat> κατά πάσα πιθανότητα τα πιο σημαντικά αλλά και τα πιο λεπτά θέματα. Η λέξη κλειδιά εδώ είναι η προσθέμενη αξία, η συνεκτικότητα, η ευελιξία και η απλότητα και ελαφρότητα του συστήματος. Δεν μπορούμε να έχουμε μια πανάκια ή ένα μοντέλο το οποίο είναι καθορισμένο από των προτέρων. Έχουν γίνει πολλές πρωτοβουλίες για να μπορέσουμε να εξευγενήσουμε λιγάκι τις βασικές ιδέες και προσεγγίσεις. Στις 27 Οκτωβρίου οργανώθηκε ένα σεμινάριο από την Βελγική Προεδρία σε στενή συνεργασία με την Φιλανδία και την Κομισιόν. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, η έννοια του κατεπήγοντος περιλαμβάνεται μέσα στη στρατηγική 2020. Ως εκ τούτου, περιλαμβάνεται και στις εξ αυτής απορρέουσες πρωτοβουλίες και επομένως η Κομισιόν προέβη σε προτάσεις φιλόδοξες, αλλά είναι περιορισμένη η πόρη μας και όσο φιλόδοξοι και να θέλουμε να είμαστε, θα πρέπει να μπορούμε να ελέγξουμε πλήρω αυτή τη διαδικασία και να αντλήσουμε συμπεράσματα εν ευθέτω χρόνο. Κλείνω κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, παρουσιάζουν την άποψη της εταιρική σχέση με καλύτερη ευκυβερνησία σε εθνικό επίπεδο. Αυτό είναι ένα ερώτημα <clears throat> το οποίο διατρέχει όλες τις σκέψεις μας σε σχέση με την ευκυβερνησία και τις εταιρικέ σχέσεις γιατί δεν υπάρχουν ήδη ρετσέτες ή έτοιμα μοντέλα και δεν υπάρχει ένα μοντέλο το οποίο τα καλύπτει όλα. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι διαφορετικέ καταστάσει από το ένα κράτο μέλο στο άλλο. Θα πρέπει να εμπλέξουμε όλου του ενδιαφερομένου, οι οποίοι μπορεί να είναι διαφορετικοί σε ένα κράτο μέλο από κάποιο άλλο. Οι εμπλεκόμενοι φορεί σε εθνικό, ευρωπαϊκό, περιφερειακό, τοπικό τομέα και ο δημόσιο και ο ιδιωτικό τομέα, όλοι πρέπει να συμμετέχουν. Κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι κοινοβουλευτικοί, είμαι πεπισμένο ότι η έρευνα και η ανάπτυξη δεν είναι απλώ επιλογή για την Ευρώπη, αλλά είναι υποχρέωση εάν θέλουμε πραγματικά με τρόπο αηφόρο να διατηρήσουμε το κοινωνικό μας υπόδειγμα και αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε την αηφορία σε επίπεδο περιβάλλοντος. Με μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν χαιρετίζω το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο σας έχει δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα θέματα αυτά και ιδίως την ε, ευκαιρία αυτή να έχω μια πρώτη παρέμβαση στη συζήτηση για το σχέδιο κοινοτομίας. Μου φαίνεται πάρα πολύ θεμελιώδης η παρέμβασή σας το σούτον μάλλον καθόσον βρισκόμαστε σε μια χρονική στιγμή που τα κρατη υποχρεωμένα να προβούν σε δύσκολες επιλογές και πρέπει να διατηρήσουμε την έρευνα και την ανάπτυξη σαν επένδυση για το μέλλον και δύναμη να σας διαβεβαιώσω ότι θα πληροφορήσω το Συμβούλιο και για το περιεχόμενο αυτής της και με φυσικά στην διάθεσή σα. Ο Μπίτι Κόφερ για διαδικαστικό θέμα. Μικρόφωνο παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ρωτήσω αν ο χρόνος ομιλίας του Συμβουλίου είναι μακρύτερος όταν συνεδριάζουμε το βράδυ. Νομίζω ότι δεν μπορεί ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου να μιλάει δύο φορές περισσότερο από ότι ο κύριος Μπαρόσο μαζί με τον κύριο Φαν Ρομπέι όταν έχουμε και άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Νομίζω ότι αυτό δεν θα πρέπει να λαμβάνει η χώρα. Μάλιστα, λέει πρόεδρος καταγράφουμε αυτό το οποίο λέτε. Σας ευχαριστούμε για την παρατήρησή σας. Έχει καταγραφεί λοιπόν. Και τώρα δίνω το λόγο στους ομιλητές συγκεκριμένων πολιτικών ομάδων και εξ του ΕΛΚ έχει καταρχήν το λόγο ο κύριος Τσουκαλάς. Θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή σας στη μεγάλη ευκαιρία που προσφέρουν οι συμπράξεις καινοτομίας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ένωσης που τόσο την έχουμε ανάγκη αλλά και στον σημαντικό κίνδυνο που υπάρχει η μη ορθή αξιοποίηση αυτού του εργαλείου να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο το χάσμα καινοτομία και έρευνας μεταξύ των κρατών μελών της ευρωπαϊκής ένωσης. αναφέρομαι συγκεκριμένα στις ε, δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σε διάφορα μέρη της Ευρώπης, αρχίζοντας από την πατρίδα μου και επισημένοντας την ίδια επισήμανση που έκανε η αξιότιμη συνάδελφος η κυρία Ματίας. Η οικονομική κατάσταση σε πάρα πολλές χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και αλλού με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαιτούν τεράστιες οριζόντιες περικοπές σε όλες τις κρατικές δαπάνες, τις δημόσιες επενδύσεις σε έρευνα περίπου να μηδενίζονται, η τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία είναι προφανές ότι κόβονται δραστικά, μιας και φαίνονται ότι αποτελούν τελευταίες προτεραιότητες στα σχέδια σωτηρίας των εθνικών κυβερνήσεων. Οι οριζόντιες περικοπές που επιβάλλονται σε αυτές τις χώρες η διαρροή εγκεφάλων που υφίστανται από εργατικό δυναμικό εξειδικευμένο που φεύγει αλλού, καθώς επίσης και οι υποχρηματοδοτήσεις πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων καθιστούν τελείως ανισοσκελές το τρίγωνο της γνώσης που πριν αναφέρατε. Αυτό το τοπίο επιδεινώνεται και από πραγματικά περιστατικά από την πραγματική επίδοση των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων για παράδειγμα η ευρώπη σύμφωνα με το times higher education που μόλις δημοσιεύτηκε προχθές έχει 82 πανεπιστήμια στα κορυφαία 200 παγκοσμίω, 80 βρίσκονται στις βόρειες χώρες και μόλις δύο τα πανεπιστήμια της Ισπανίας βρίσκονται στο Νότο. Θέλω να ρωτήσω την Κομισιόν, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κοινοβούλιο ή όποιον μπορεί πώς σκοπεύουμε να αντιμετωπίσουμε το διαφαινόμενο χάσμα ανάμεσα στην καινοτομική Βόρεια Ευρώπη και τον Ευρωπαϊκό Νότο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Σας παρακαλώ να παραμένετε στον χρόνο αγόρευσή σας. Και τώρα δίνω το λόγο στην κυρία Ριέρα μαδουρέλα Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι γεγονός ότι είναι πολύ επιτυχημένη η πρόταση της Κομισιόν για την καιροτομία μαζί με την πρότασή της για τη βιομηχανική πολιτική. Για να μπορέσουμε να έχουμε οικονομική ανάπτυξη με ανταγωνιστικότητα και απασχόληση, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποχρεωμένη να βελτιώσει την ικανότητά της να καινοτομεί. Η πολιτική μας ομάδα έχει υποστηρίξει και τις δύο αυτές και ω συντονίστρια εγώ είμαι σίγουρη ότι με τη συνεργασία όλων μας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορέσει να βρει λύσεις για αυτές τις νέες προκλήσεις. Λύσεις που δίνουν μια ισορροπία μεταξύ του οικονομικού, του κοινωνικού και του περιβαλλοντικού για να προχωρήσουμε προ μια Ευρώπη πιο ευφυά και πράσινη με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Το ψήφισμά μας λοιπόν τονίζει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας κατάλογος θεμάτων κατά προτεραιότητα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της συνεργασίας για την καινοτομία, τονίζοντας ότι η επιτυχία στους τομείς αυτούς θα εξαρτάται από την ικανότητά μας να εμπλέξουμε <clears throat> σε αυτά τα εγχειρήματα τόσο τις καινοτόμες επιχειρήσεις όσο και τα πανεπιστήμια και τα κέντρα έρευνας και καινοτομίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα εξ ονόματος των συντηρητικών, της ομάδας των συντηρητικών, ο κύριος Ζομπρό. Πρόεδρε κύριε και κύριοι, η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει την καινοτομία γιατί αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσει την τωρινή κρίση. Ένα δε στοιχείο κλειδί για να υπάρξουν τέτοιες αλλαγές θα ήταν να αυξηθούν οι επενδύσεις στον τομέα της καινοτομίας με ευέλικτη νομοθεσία που να προωθεί τις επιχειρήσεις, να είναι σε θέση να παίρνουν πιο εύκολα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και copyright δικαιώματα. Όσο για την ε, χρηματοδότηση πολιετών προγραμμάτων, εκεί μπορεί να υπάρξουν προβλήματα, διότι μπορεί να μην αρκεί ο προπολογισμό και χρειάζονται οι επιχειρήσεις να κάνουν μαζικές επενδύσεις δικές τους. Αυτό είναι άσκημο νέο για τους επενδυτές στην Ανατολή, στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που δεν μπορεί να μην έχουν πρόσβαση σε ενωσιακή χρηματοδότηση. Αυτό φαίνεται καθαρά από πολλά παραδείγματα και σημαίνει ότι ορισμένες εταιρείες σε ορισμένα μέρη της Ευρώπης μπορούν να κάνουν επένδυση στην έρευνα και άλλες όχι. Αυτό δημιουργεί χάσμα. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω τι μπορείτε να κάνει η Κομισιόν για να γεφυρωθεί το χάσμα αυτό. Ευχαριστούμε. Και τώρα μονομενή βουλευτέ. Πρώτα ο κύριος Βίνκλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι με την πρόταση για την καινοτομία η Ευρωπαϊκή, Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια κατά την άποψή μου σωστή κατεύθυνση. Και με την ε, πρότασή της, της ε, του Σεπτεμβρίου του 2010 χαράσει έναν δρόμο τον οποίο τον ενέκρινε η Επιτροπή Βιομηχανία και Έρευνα, γιατί με τον τρόπο αυτό θεωρούμε ότι μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει καλύτερα το δυναμικό τη στον τομέα τη έρευνα και τη ανάπτυξη και να μπορέσει να ανταγωνιστεί χώρε όπω οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ιαπωνία, όπω και αναδυόμενε οικονομίε όπω η Κίνα. Αλλά θα έχουμε επιτυχία στον τομέα αυτό μονάχα όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη και με τι περιφέρειε τη Ευρώπη. Γι' αυτό <clears throat> προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη λεγόμενη εταιρική σχέση για την καινοτομία που ε, θα πρέπει να αναλυθεί και κατατομής με τον κατάλληλο τρόπο. Νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό δημιουργείται και πάλι μια διτή ε, δομή και ούτως ή άλλως η έννοια της εταιρική σχέσης δεν είναι ακόμα σαφής και το Συμβούλιο δεν κατάφερε με τις δικές του προσπάθειες να τη διαλευκάνει περισσότερο. Η ιδέα της εταιρική σχέσης με την, για την καινοτομία μοιάζει πάρα πολύ με προηγούμενα όργανα που υπήρχαν στο παρελθόν, όπως είναι οι τεχνολογικές πλατφόρμες στα πλαίσια των προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης. Θέλω να υπενθυμίσω ότι θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες προσπάθειες ώστε να εξασφαλίσουμε τη συνέργεια μεταξύ των εμπλεκομένων, να χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα αυτή τη συνέργεια και να μπορέσει να διατηρηθεί ένα συνεκτικό πλαίσιο για την εκτέλεση αυτών των ενεργειών. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κουρία Ντεκάμπους έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Χαιρετίζουμε τις προσπάθειες Ευρωπαϊκής Επιτροπής ούτως ώστε να ανεδειχθεί σε ύψιστη πολιτική προτεραιότητα η καινοτομία και η έρευνα. Θέλουμε μια πλήρη πολιτική ούτως ώστε το ευρωπαϊκό σύστημα να είναι πιο αποτελεσματικό και να εξυπηρετεί μια βιώσιμη οικονομία. Οι ευρωπαϊκές εταιρικές σχέσεις για την καινοτομία είναι ένα χρήσιμο εργαλείο και οι προκλήσεις ε, που οργανώνονται νομίζω δεν πρέπει να είναι αμφιλεγόμενες. Ε, ε, βεβαίως θα πρέπει να ορίσουμε τις θεματικές προτεραιότητες και να δούμε και τους υποτομείς μέσα σε κάθε θεματική ενότητα ούτω ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν όλοι οι εταίροι. Ποιο είναι ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, των κρατών μελών, των περιφερειών, και πώς θα εξασφαλίσουμε τη λογοδοσία με αυτό τον περίπλοκο μηχανισμό και ποια η δημοσιονομική, ε, ο δημοσιονομικός χαρακτήρας αυτών των πρωτοβουλίων ε, χρειάζεται αριστεία στην υλοποίηση και εφόσον δεν έχουμε ακόμη εγγυήσεις ε, για αυτά τα πιλωτικά προγράμματα της πρώτης εταιρικής σχέσης νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Γκουτιέρες Κορτίνες. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να τονίσουμε την αξία της καινοτομίας. Αλλά μιλάμε για κάτι που πραγματικά δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι. Είναι μια πρωτοβουλία για την οποία συζητούμε χωρίς να ξέρουμε ποιο είναι το περιεχόμενο. Ούτε η φόρμουλα που ακολουθείται, ούτε το υπόδειγμα που διατρέχει αυτή την πρωτοβουλία. Εγώ τονίζω ότι αν θέλουμε να είμαστε αποδοτικοί και αποτελεσματικοί, θα πρέπει να δούμε τα αποτελέσματα των προηγουμένων πρωτοβουλειών μας τι έχει γίνει με τις εταιρικές σχέσεις, τι έχει γίνει με τις ερευνητικές πλατφόρμες. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα θέματα με πραγματικά αντικειμενικό τρόπο, με εξωτερικές ε, αξιολογήσεις. Είδαμε σε πολλές περιπτώσεις ότι όλη η ερεύνα κυριαρχείται και καταδυναστεύεται από τις μεγάλες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Εγώ θα πρότεινα να υπάρχουν κάποιες φόρμουλες και κάποιες πολιτικές καινοτομίες που να ενισχύουν και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να μπουν στο χώρο της αγοράς. Να έχουμε ενδιαμέσους οι οποίοι θα βοηθήσουν αυτές τις εταιρείε να συμμετέχουν στα σχέδια αυτά. Δεν μπορούμε να τις κρατάμε πάντα στο περιθώριο. Επίσης θα πρέπει να σκεφτούμε και καινοτομία σε επίπεδο διαχείρισης και ελέγχου της καινοτομία. Γιατί θα πρέπει να ακολουθεί η διοίκηση και οι δικαιωτικέ δομέ, να ακολουθούν την αγορά που είναι πολύ πιο γρήγορε από τι ίδιε τι δομέ αυτέ. Επομένω, θα πρέπει να έχουμε δομέ οι οποίε είναι κατάλληλε για τη διαχείριση των καινοτομιών και που θα βοηθούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπουν στο χώρο αυτό της καινοτομίας το οποίο είναι πιο σημαντικό και επίσης να μπορούμε να τις βοηθούμε να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους που δεν πρέπει να τους φέρει μονάχα φορολογούμενος. Η κυρία Τσίκαου έχει το λόγο τώρα. Ένα λεπτό. Σίλβια Αδριάννα Τσικάου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η βασική διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τονίζει ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στην πολιτιστική ζωή της κοινότητάς του, στην καλλιτεχνική ζωή και να απολαμβάνει των επιστημονικών προόδων. Πρέπει λοιπόν η καινοτομία να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα μεταξύ των οποίων τις κλιματολογικές αλλαγές, την έλλειψη ορισμένων πρώτων υλών κλπ. Για να μπορέσει η Ένωση να αναπτύξει τη δυνατότητα καινοτομία της που είναι τόσο ουσιώδης για την ανταγωνιστικότητά της πρέπει να καταφέρουμε να συνδυάσουμε τη βιομηχανική πολιτική με πολιτική καινοτομία, να αναπτύξουμε την παραγωγικότητά μας και την, να αυξήσουμε τις θέσεις των αριθμό των θέσεων εργασίας. Όλα αυτά βέβαια βασίζονται στην καινοτομία η οποία με τη σειρά της εξαρτάται από την διάδοση των επιστημονικών γνώσεων. Χρειάζεται λοιπόν μια νέου τύπου εταιρική σχέση που να διευκολύνει την παιδεία για να υπάρξει μεγαλύτερη επιστημονική πρόοδος. Ευχαριστούμε κύριε Τζουκάου. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Χιούμπνερ για 1,5 ολόκληρο λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι. Τα τελευταία χρόνια έχουν υποθεί πολλά για την καινοτομία και έχει γίνει μια, ένα εμβληματικό μέσο και θεωρείται πανάκια. Ε, υπάρχουν σοβαρές προσδοκίες και πρέπει να έχουμε τα κατάλληλα αποτελέσματα και κυρίως αυτή τη χρονική στιγμή πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Ε, η καινοτομία μπορεί να έχει κρίσιμο ρόλο για την τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας αλλά για να γίνει αυτό θέλουμε ε, μια κοινή ε, προσπάθεια δημόσιο ιδιωτικού τομέα, τόσο ώστε να ισχύσουν καλύτερε προποθέσει πλαίσιο, πρόσβαση στη χρηματοδότηση, επανεστιασμό των πολιτικών. Αλλά αυτό που μα χρειάζεται περισσότερο είναι ο χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει να κινηθούμε γρηγορότερα, να περάσουμε από τα λόγια στι πράξει, να καταργήσουμε του ανασχετικού παράγοντε και πρώτα απ' όλα να σχεδιάσουμε νέα εργαλεία πολιτικής που να είναι αποτελεσματικά. Οι εταιρικέ σχέσεις καινοτομία μπορεί να ε, συνιστούν ένα καλό εργαλείο και να οδηγήσουν σε αριστεία. Κατά τη γνώμη μου είναι κατεπήγον το ζήτημα και η προσέγγιση μας θα πρέπει να είναι ε, βλέποντας και κάνοντας. Έτσι μόνο θα μάθουμε και υπάρχουν εξάλλου πρακτικές στην Ευρώπη. Ε, και κανονικά οι περιφέρειες παίζουν ρόλο κλειδί στις περιφέρειες ε, και τι μπορούμε να κάνουμε να επισπεύσουμε την, ε, το δρόμο προς μια ε, καινοτόμα οικονομία ενισχύοντας τις επενδύσεις με 85 δις ευρώ και να αναλάβουμε τις κατάλληλες δεσμεύσεις μετά το 2013 για την έξυπνη ανάπτυξη. Και έτσι θα είναι επωφελής οι εξελίξεις για όλες τις χώρες και για όλες τις περιφέρειες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα στον συνάδελφό μου τον κύριο Μπαλτσίτης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η πολιτική καινοτομία και η τεχνολογική επιτυχία χρειάζονται διευκολυντικούς παράγοντες για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της Ευρώπη 2020 και σε μια Ευρώπη η οποία είναι ανταγωνιστική. Εδώ παίζει ιδιαίτερο ρόλο και η αποδοτικότητα της ε, χρήσης ενέργειας, οι καθαρές τεχνολογίες, ο μετριασμός των συνεπειών τη κλιματική αλλαγή. Όλα αυτά εξαρτώνται από την αποτελεσματικότητα τη πολιτική καινοτομία στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια ολοκληρωμένη πολιτική, κάτι το οποίο μπορεί να επιτευχθεί μονάχα αν έχουμε αποτελεσματική συνεργασία και διαχείριση σε τοπικό, περιφερειακό, ευρωπαϊκό εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής για την καινοτομία με εταιρική σχέση είναι μια θαυμάσια πρωτοβουλία που θα μας επιτρέψει να έχουμε καλύτερο αποτελέσμα στον τομέα της ανταγωνιστικότητας και θα δώσει μεγαλύτερη πρόοδο στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ, Λέω ο Ο κύριος Πυρίλο, ο Μάριο Πυρίλο, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τη στιγμή που υπάρχουν προγράμματα λιτότητος σε πάρα πολλά κράτη-μέλη φαίνεται ότι η καινοτομία είναι το κλειδί που θα επιτρέψει την, στην Ευρώπη να βγει από την κρίση. Είναι πάρα πολλές, περι... πολλές εφευρέσεις οι οποίες άλλαξαν την μορφή του κόσμου έχουν ξεκινήσει από τη δική μας Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Το μεγάλο πνευματικό κεφάλαιο που έχει η Ευρώπη και στον επιστημονικό τομέα θα πρέπει να τύχει εκμετάλλευση με κοινέ δράσει των κρατών μελών και τη Ευρωπαϊκή Ένωση που θα αποφεύγουν τι αλληλοεπικαλύψει και θα βελτιστοποιούν τι ε, επενδύσει. Πρέπει να έχουμε μια πιο συντονισμένη και πιο στρατηγική διαδικασία επενδύσεων. Γι' αυτό οι εταιρικέ σχέσει στον τεχνολογικό τομέα είναι πάρα πολύ σημαντικέ. Θα ήθελα να ρωτήσω το Συμβούλιο με ποιο τρόπο θα κάνει πιο δυναμικές αυτές τις εταιρικέ σχέσεις και πώς θα μπορέσει να μεταλαμπαδεύσει τα αποτελέσματα αυτών των εταιρικών σχέσεων στην πραγματική οικονομία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πυρίλου. Μας φέρνει αυτό στο τέλος των παρεμβάσεων των βουλευτών από τις πολιτικές ομάδες και μεμονωμένα. Και τώρα αρχίζει η διαδικασία Catch the Eye. Ο κύριος Κέλλη έχει πρώτος το λόγο. Σον Κέλλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χωρίς καμιά αμφιβολία είναι μεγάλη η πρόκληση αυτή. Και είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να βρούμε νέους τρόπους να, δια... να διαπραγματευτούμε και να λύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Εδώ βλέπετε το βαρόμετρο της καινοτομίας που έχει και μία επισκόπηση όλων των εμπλεκομένων στον τομέα αυτό. 90% τόνισαν ότι η καινοτομία θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη της οικονομίας και 83% αυτών που απάντησαν θεωρούν ότι οι εταιρικέ σχέσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι απαραίτητες για μια πιο καινοτόμα Ευρώπη. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ καλό δεκτή η σημερινή συζήτηση. Σήμερα είχα διοργανώσει ένα γεύμα με εκπροσώπους του Συμβουλίου και της Κομισιόν μαζί και με ευρωβουλευτέ για το θέμα αυτό των εταιρικών σχέσεων για την καινοτομία. Το κλειδί του μέλλοντο, αν θέλουμε να πετύχουμε το στόχο τη Ευρώπη του 2020, είναι 3% του ΑΕΠ για την έρευνα και την ανάπτυξη και επίση διατήρηση του ανθρώπινου κεφαλαίου που είναι απαραίτητο. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ιωάν Έντσου, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να χαιρετήσω τις προτάσεις της Κομισιόν για, την, για το πρώτο αυτό πρόγραμμα εταιρικής σχέσης για την καινοτομία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει πιο ενεργά να δραστηριοποιηθεί στον τομέα των επενδύσεων εξισορρόπησης μεταξύ της συνδιαχείρισης των κρατών μελών και της έρευνας. Πρέπει να δώσουμε την προσοχή που αρμόζει σε αυτό το θέμα και πρέπει να επιδείξουμε μεγάλη συνέπεια. Οι δημόσιες επενδύσεις των χωρών μελών και οι ιδιωτικές τιάφτες πρέπει να συνδυαστούν. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Έντσιου, στην κυρία Έντζιου. Αμάν. Σας ευχαριστώ η καινοτομία είναι κάτι που έχει γίνει πια σύνθημα της μόδας. Πρέπει όμως να ομολογήσουμε ότι ναι, δεν πρόκειται δεν πρόκειται λέγω να καταλήξει πουθενά σύντομα διότι η ανάπτυξη προϊόντων χρειάζεται χρόνια ολόκληρα και το κόστος της ανάπτυξης προϊόντων επιβαρύνεται συνεχώς. Πράγμα που σημαίνει ότι στην Ευρώπη πρέπει να κάνουμε σοβαρές επενδύσεις σε κοινή έρευνα και με βάση την εσωτερική αγορά. Δεν πρέπει να αναμένουμε μόνο ενωσιακές λύσεις. Η καινοτομία θα φέρει τους καρπούς της εν καιρό το δέοντι. Αλλά δεν πρόκειται για πανάκια. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ιλντα Φιγκερέιντο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πρόκληση ποια είναι αυτή η πρωτοβουλία, δηλαδή ε, η Ευρώπη της καινοτομίας, είναι εμπληματική, αλλά να μην μείνουμε σε αυτό, να μην είναι ένα λάβαρο, αλλά να ενσωματωθεί σε μια πραγματική αναπτυξιακή πολιτική, πολιτική κοινωνικής προοδού, όπου η καινοτομία θα είναι ένα σημαντικό εργαλείο. Αλλά για να, ε, για να είναι αποτελεσματικό αυτό το εργαλείο θα πρέπει να έχουμε τις απαιτούμενες δημόσιες πολιτικές. Το πιλωτικό πρόγραμμα για, σε αυτό το τομέα είναι ήδη υποδειγματικό. Επίσης, θα έχουμε σημαντικά αποτελέσματα εάν συνοδευτούν τα μέτρα από δημόσιες πολιτικές, ούτως ώστε να προσφέρονται ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες, να υπάρχει ε, κοινωνική προστασία, εξοπλισμός και υποστήριξη προς τους ηλικιωμένους για μια ε, αξιοπρεπή γύρανση. Ας μην παραδοθούμε στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητες που πλήττουν την ποιότητα ζωής των πληθυσμών ε, πληθυσμιακών ομάδων, κυρίως των ηλικιωμένων. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτω ώστε αυτή η πρωτοβουλία να μην μείνει κενό γράμμα. Ε, τελευταίος, Αλεξίσου, σημαντικός ο κύριος Ματούλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η οικονομία η οποία είναι αηφόρος και ευφύης για την επίτευξη των στόχων του 2020 είναι απαραίτητη. Και αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα μόνο με την υποστήριξη της καινοτομία και της έρευνας. Πρέπει να προωθήσουμε λοιπόν ε, όλες τις μεθόδους όπως η διαμεθοριακή συνεργασία μεταξύ κράτων μερών για να ευδοκιμήσει αυτή η στρατηγική. Πρέπει να ξεκινήσουμε εκ των κάτω προς τα άνω. Οι λύσεις θα προέλθουν από την ε, καινοτομία στι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν καταρχήν μεγάλες δυσκολίες. Για το λόγο αυτό οι περιφερειακές αρχές θα πρέπει να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο για να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν αυτούς τους υπνώτοντες καινοτόμους όπως έχουμε χαρακτηριστεί μέσα στα πλαίσια της πολιτικής καινοτομία. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βελτιώσουμε την καινοτομία, να ενισχύσουμε τις σχέσεις μεταξύ των αποδεκτών των κονδυλίων και των καινοτόμων και να δημιουργηθούν εταιρικέ σχέσει προ την κατεύθυνση αυτή. Με την ευκαιρία τη ε, επίσκεψη που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα παρουσιάστηκαν ε, διάφορες πρωτοβουλίες από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης από τις οποίες προέρχομαι και εγώ και νομίζω ότι αυτές οι σχέσεις μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος και τώρα για να κλείσουμε δίνω το λόγο στον Υπουργό Σερέξ. Σας παρακαλούμε κάντε ε, μια σύνοψη της συζήτησης. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Κοινοβούλιο για το ενδιαφέρον που έδειξε για το φάκελο της καινοτομίας. Αυτή η υποστήριξη είναι πραγματικά απαραίτητη για να υλοποιήσουμε αμελητή, κατεπηγόντως, ε, ε, το σχέδιο για την καινοτομία και για να ανταποκριθούμε στις εσωτερικές προκλήσεις αλλά και για να ε, ευελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας ε, στις εξωτερικές μας σχέσεις. Μου είπατε να είμαι σύντομος θα είμαι. Ε, δεν είχαμε και χρόνο στη διάθεσή μας. Στις 6 Οκτωβρίου υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρότασή της και τώρα εμείς προετοιμάζουμε τα συμπεράσματα για το Συμβούλιο της 26 Νοεμβρίου. Όλοι γνωρίζουν ότι η έρευνα και η καινοτομία είναι απαραίτητα απαραίτητα για να εξέλθουμε από την κρίση. Ε, για την επιλογή των εταιρικών ε, σχέσεων ε, τώρα, τόνισα τη σημασία του πρώτου θέματος που θα μας οδηγήσει στο πιλωτικό πρόγραμμα, δηλαδή να δούμε κατά πόσο είναι εφικτό αυτό το μοντέλο και το πρώτο αυτό πιλωτικό πρόγραμμα νομίζω ε, μπορεί να οδηγήσει σε συσπήρωση των ε, ενδιαφερομένων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερθηκε και σε άλλες 12 θεματικές ενότητες και το Συμβούλιο θεωρεί ότι το σημαντικό είναι να έχουμε μία αύξουσα ε, πορεία, αύξηση ε, του αριθμού των προγραμμάτων και κυρίως να αποφύγουμε τις ε, επικαλύψεις και να δημιουργήσουμε επιπρόσθετες δυσκολίες με επιπρόσθετα προγράμματα. Όχι. Αυτό αντιβαίνει στο στόχο μας που είναι η απλούστευση μεταξύ άλλων. Για το δημοσιονομικό πρόβλημα τώρα. Ε, γνωρίζουμε την πίεση που ασκείται σε όλους τους προϋπολογισμούς και όπως ακούστηκε και προηγουμένως θεωρώ ότι η αριστεία πρέπει να είναι ένας κοινό ε, στόχος. Αυτό δε θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη στο ε, συντονισμό της δράσης διαφόρων μέσων που διαθέτουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως δηλαδή ανάμεσα στο πρόγραμμα πλαίσιο και στα διαρθρωτικά ταμεία. Στο Συμβούλιο Ε, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε όλους ιδιαίτερως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί στο παρελθόν δεν είχαν επαρκή πρόσβαση στο προηγούμενο πρόγραμμα πλαίσιο και γι' αυτό εμείς εμένουμε στη σημασία της απλούστευσης και της ευκολότερης πρόσβασης στη χρηματοδότηση και στους όρους πλαίσιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε Υπουργέ. Και έτσι φτάνουμε στο πέρας της συζήτησης σε αυτού του σημείου. Έχουμε καθυστερήσει.